δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα υπάρξουν οι παναχωρήσεις στην πολιτική γραμμή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκάλου. Ο κύριος Φόμποντα για ένα μισή λεπτό έχει το λόγο.